Colleghe colleghi, prendete posto. Καθίστε σας παρακαλώ συνάδελφοι. Il processo verbale. Τα πρακτικά, τα συνοπτικά πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν στη θεσινή συνεδρίαση διατίθενται. Παρατηρήσεις έχετε επί των πρακτικών. Εγκρίνονται λοιπόν τα συνοπτικά πρακτικά. Έχεις δει το λόγο. Η κυρία Ντουράν, της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι στα έδρανά σας θα βρείτε ένα φάκελο που αφορά το βραβείο Λουξ Όπω γνωρίζετε είναι ένα κινηματογραφικό βραβείο το οποίο θα απονείμετε εσείς. Και θα ήθελα να σα θυμίσω, σας παρακαλώ, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι μπορείτε να ψηφίσετε. Οφείλετε να ψηφίσετε για να επιλέξετε ένα από τα τρία φίλμια από τις τρεις ταινίε που διαγωνίζετε. Έχετε λοιπόν αυτό το φάκελο και ένα DVD της ταινία που κέρδισε το 2007 και μεταφράστηκε σε 27 γλώσσες, συγγνώμη, 23 διορθώνει ομιλήτρια, συν 7, για να μπορούν όλοι οι Ευρωπαίοι να βλέπουν τις ταινίε αυτές. Λοιπόν, σας ζητώ τα εξής τρία. Πρώτον, να πάτε να δείτε τις ταινίε που διαγωνίζονται. Σας παρακαλώ πολύ. Ah, να πάτε να δείτε τις ταινίε. Να ψηφίσετε, είναι πολύ εύκολο να ψηφίσετε. Γράφει στο φάκελο τη διαδικασία, μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά ε, ή και στην τηλεόρασή σας να δείτε την ταινία στο κανάλι 77. Δείτε παρακαλώ τις ταινίε, είναι ωραία έργα κινηματογραφικά, ε, προάγουν τις ευρωπαϊκές αξίες, μπορείτε να ψηφίσετε ένα, δύο ή τρία. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να ψηφίσει Πολλοί βουλευτέ παρακαλώ να συμμετέχετε μαζικά. Είναι μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Είναι μια πρωτοβουλία των πολιτών που προάγει τι ευρωπαϊκέ αξίε και του ευρωπαίου σκηνοθέτε. Λοιπόν, ε, το μπαλάκι τώρα είναι σε εσά. Έχετε μια εβδομάδα για να ψηφίσετε. Υπολογίζω στη συνεργασία σα και σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού, την κυρία Τόρι Πακ, η οποία πάρα πολύ ε, βοήθησε σε αυτή την προσπάθεια και εκείνη και εγώ σας ζητούμε μαζικά να ψηφίσετε σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ντουράν. Ωραία, μας δώσατε και ε, τροφή για το Σαββατοκύριακο. Και με πολύ μεγάλη προσοχή θα κάνουμε αυτό που μα είπατε. Περνάμε τώρα στη μερίσια διάταξη στις ψηφοφορίες. Ψηφίζουμε την έκθεση κυρία Φαγιών για τον κατάλογο των τρίτων χωρών, των οποίων οι πολίτες θα πρέπει να έχουν θεώρηση ε, όταν περνούν τα εξωτερικά σύνορα ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση